Ξεκινάμε το ψήφισμα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην, Κρεμή, στην Κρυμαία και ιδιαίτερα την κατάσταση των Τατάρων. Παράγραφη 7, προφορική τροπολογία του κυρίου Πλένκοβιτς. Κύριε Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την ε, προφορική τροπολογία για την παράγραφο 7, είναι τεχνικό ζήτημα, κάτι το οποίο συμφωνήσαμε στις διαπραγματεύσεις και είναι κάτι το, στο οποίο συμφώνησαν όλες οι ομάδες. Σας ευχαριστώ. Άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιδη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε σε κοινό έτοιμο από έξι ομάδες που αφορά την ε, περίπτωση Ραμαντάν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η παραγραφός 3 εκτιμώντας α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας όμικρον υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ψήσιμο στο σύνολό του υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κοινό έτοιμο ψήσιμο από έξι ομάδες. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. απολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολο του υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Ακολουθεί. Το ψήφισμα της Επιτροπής Εξωτερικών παράγραφος 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Παράγραφος 18, ε, μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγραφος 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή παράγραφος 30 αρχικό κείμενο μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Το ψήσιμο στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Δεκτό. Και πάλι από την Επιτροπή Εξωτερικών αφορά το κοσυφοπέδιο, Το 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Επί της διαδικασίας η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Για την επόμενη τροπολογία του ΕΛΚ, για την οποία η συμβαστική λύση πριν την ψηφοφορία, ήθελα να ευχαριστήσω τον σκιώδη συγγητή του ΕΛΚ, που δέχτηκε να αποσύρει τη δική του τροπολογία περιθμών 8 και να συμφωνήσει επί του κειμένου καλεί την ε, ε, επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ναι, αυτό το τμήμα να παραμείνει. Αυτή είναι λοιπόν η δική μου συμβαστική λύση με τη στήριξη του ΕΛΚ και θα παρακαλέσω όλους τους κοιότητες εισηγητές να συμφωνήσουν. Δεν είχαμε χρόνο να το συμφωνήσουμε νωρίτερα, ε, διότι ήταν τελευταία στιγμή η λύση που εξευρέθη. Θα σας παρακαλέσω να το δεχτείτε. Gibt Δεν βλέπω. Ψηφίζουμε λοιπόν την παραγραφό 6 αρχικό κείμενο. Αντιρρήσεις. Ναι, παρακαλώ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους του ΕΛΚ θα συμφωνήσω με όσα είπε η κυρία Λαγνάτσεκ. Ψηφίζουμε λοιπόν το αρχικό κείμενο της παραγράφου 6 χωρίς το κομμάτι που μας είπε η κυρία Λούνατσικ λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτό παράγραφος ε, τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 10 σε 3 μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος τρίτο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 14 αρχικό κείμενο σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παράγραφος 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Παράγραφος 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Παράγραφος 23 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 με ονομαστική ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Θα το Δούμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για τροπολογία 3. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα πέντε ομάδων που αφορά την κατάσταση στη Λιβύη. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παραγραφός 6, 2 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό μέρο δεύτερο σε ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 11 αρχικό κείμενο. Μέρος πρώτο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Μέρος δεύτερο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Δεκτό. Τροπολογία 6 πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12. Αρχικό κείμενο μοναστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Δεκτό. Τροπολογία 1. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας ένα μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Εκτιμώντας Β, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εφεκτό. Έχουμε τώρα το ψήφισμα που αφορά την ισιωτικότητα. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 1. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές δεκτό πρόταση ψηφίσματος από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον τόπο των ΟΤΑ στα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Παράγραφος 2 του αρχικού κειμένου μέρος 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα που αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση στην Έχουμε πρόταση ψηφίσματος. Πρώτα του ECR. Υπέρ. Κύριε Πρέντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι διαπραγματευτέ από τι διάφορε πολιτικέ ομάδε δέχτηκαν την αναβολή τη ψηφοφορία αυτή για την επόμενη σύνοδο. Σα ευχαριστώ, ελπίζω να το δεχτείτε. Θέλει κάποιο να τοποθετηθεί υπέρ. Υπέρ. Υπέρ. Κύριε Χάουιτ. Ευχαριστώ. Προείδρευσα στις δημοτεύσεις για το ψήφισμα αυτό. Κατόπιν αιτήματος της ομάδας μου και στη συζήτηση με τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και το ΕΛΚ συμφωνούμε με την αναβολή. Δύο εβδομάδες είναι μόνον. Αν και υπάρχει ανθρώπινη ανάγκη, ανθρωπιστική ανάγκη κατεπίγουσα εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε άμεσα. Πιστεύουμε ότι η επιρροή μας θα αυξηθεί εφόσον είναι ισχυρή αυτή η ψηφοφορία. Η αναβολή όμως θα μπορούσε να ήταν για κάποιους ε, δόλιο σχεδίο για να υπονομευθεί η ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου. Στην αρχή, στο αρχικό κείμενο το ΕΛΚ δεν μπορούσε να προσυπογράψει στο αρχικό κείμενο. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε αντίρρηση για την ώρα, αλλά ο καλύτερος τρόπος να ασκήσουμε επιρροή είναι ένα ισχυρό ψήφισμα. Κατά ο κύριος Σμιθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν συμφωνούμε με αυτή την αναβολή, διότι η κατάσταση στην Ιεμένη είναι πολύ σοβαρή. Το κείμενο αυτό το επεξεργαζόμαστε εδώ και καιρό και υπάρχει η πλειοψηφία. Ε, ισχυρή και προοδευτική θέση και τοποθέτηση για την σύγκρουση αυτή, την αιματηρή αυτή χρονοπραξία ε, και αντιπαράθεση υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα λόγο στο ψήφισμα αυτό να ψηφιστεί τώρα. Είναι ήδη πολύ καλό. Υπάρχει πλειοψηφία εδώ για να έχουμε μια θέση που μα ε, ε, εξυπηρετεί. Οπότε δεν βρίσκω κανένα λόγο να υπάρξει ένα πολύ ευχαριστώ. Ψηφίζουμε το αίτημα αναβολή. Ποιο είναι είναι υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Αναβάλλεται λοιπόν το αντικείμενο της ψηφοφορίας. Περνάμε σε κοινή πρόταση ψηφίσματος 6 ομάδων όσον αφορά τις συστηματικές δολοφονίες το Ισλαμικό κράτος. Το τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παραγραφός 10. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ναι Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές δεκτό Περνάμε τώρα στις ε, επεξηγήσεις ψήφου. Και ο συνήθως ε, θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους να εγκαταλείψουν την αίθουσα ησύχως.